δώσατε, όλες οι απα... για τις απαντήσεις, για τη ζωηρή συζήτηση και είναι πολύ σημαντικό να δίδονται ευρωπαϊκές απαντήσεις στην τραγωδία της Ιαπωνίας. Ευχαριστώ εκ νέου κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους επιτρόπους που είναι παρόντες εδώ. Ευχαριστώ. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Συντονισμού των Εθνικών Στρατηγικών για την ένταξη των τσιγκάνων. Και δίνω το λόγο αμέσως τώρα στην Επίτροπο την κυρία Ρέντινγκ. Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μαζί με τον Λάσλο Άντορ, τον συνάδελφό μου, θα σας παρουσιάσουμε την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβολή ενός ενωσιακού πλαισίου για τον συντονισμό των εθνικών στρατηγικών ένταξη των Ρωμά. Αυτό το πλαίσιο έρχεται σε μια στιγμή όπου η κατάσταση των Ρωμά έχει έρθει στο επίκεντρο της προσοχής στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει στα κράτη-μέλη ένα φάσμα νομικών, μάλλον εργαλείων πολιτικής, και νομικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και υπάρχει και μια νομική βάση για την μη διακριτική μεταχείριση και την ελευθερία μετακίνησης ή τη στρατηγική διεύρυνση. Βέβαια, είναι σαφές ότι στο επίπεδο το κοινωνικό και το οικονομικό η περιθεριοποίηση των Ρωμά παραμένει. Και αυτό δεν είναι αποδεκτό. Ούτε μπορεί να συνεχιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την υποστήριξη όλου του πολιτικού φάσματος και θέλω αυτό να το τονίσω επέστησε την προσοχή μας ε, στον ανάγκη κατεπηγόντως να προωθήσουμε την ένταξη των Ρώμα μέσω ενός ε, ψηφίσματος που ενέκρινε πρόσφατα για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τους Ρωμά. Σήμερα ήταν η κυρία Ζαρόκα, την οποία θέλω να την ευχαριστήσω για το εξαιρετικό της έργο. Χρειάζεται λοιπόν αποφασιστική δράση και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κλιμακώσουμε τις προσπάθειές μας για την, ε, να πάψει η διακριτική μεταχείριση κατά των Ρωμά, ώστε να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλο Ευρωπαίο πολίτη, διότι και αυτοί είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Και όταν το λέω αυτό, φυσικά και εννοώ μία αμφίδρομη διαδικασία που απαιτεί αλλαγή νοτροπίας, αλλαγή θεώρησης και αντιλήψεων και αυτό αφορά και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα μέλη της κοινότητας των Ρωμά. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός και εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών. Καθώς επίσης και μια στρατηγική κοινή προσέγγιση. Γνωρίζουμε ότι η πρωταρχική ευθύνη για την ένταξη των Ρωμά είναι, στα ευθύνη των κρατών μελών. Αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα όμως ότι η κατάσταση των Ρωμά ποικίλει, ποικίλει σημαντικά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρουσιάσει ένα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, τα κράτη-μέλη δράση αναλογικά με τη δική τους, ε, την έκταση του προβλήματος στη δική τους χώρα. Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο ε, κάποιες ε, διαβουλεύσεις και κάποιες έρευνες και είδαμε ότι πολλές φορές δεν γίνονται πολλά. Τα 26,5 δις ευρώ που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων δεν αξιοποιούνται με τον τρόπο που θα έπρεπε και μόνο 100 εκατομμύρια ανατέθηκαν σε συγκεκριμένες δράσεις υπέρ των Ρωμά και μόνο μάλλον και το 70% των μέσων για την παροχή τεχνικής βοήθειας τα οποία θα χρειαστούν στα περισσότερα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιήθηκαν. Επομένως, τα μέχρι τώρα υφιστάμενα μέτρα δεν είναι επαρκή. Καιρός είναι λοιπόν πια να εξασφαλίσουμε ότι οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές θα επικεντρωθούν σε ανάγκες των Ρωμά με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο. Στο πλαίσιο λοιπόν που προτείνουμε επικεντρωνόμεθα σε τέσσερα βασικά θέματα. Παιδεία, απασχόληση, υγεία, στέγαση. Θέλουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα 27 κράτη-μέλη να δεσμευθούν για τη γεφύρωση του χάσματος, να επικεντρωθούν στους κοινούς στόχους αυτούς τους τέσσερις τομείς, με στοχευμένες δράσεις, με επαρκείς πόρους για να επιτύχουν αυτοί οι στόχοι. Θέλουμε όλα τα κράτη-μέλη να εντάξουν τους στόχους αυτούς ε, στην φυστάμενη στρατηγική ε, που έχουν, αν έχουν, για τους Ρώμα ή να αναπτύξουν στρατηγική για τους Ρώμα, εάν δεν έχουν, για την περίοδο μέχρι το 2020 και προκειμένου να επαληθεύσουμε κατά πόσον οι προσπάθειες ε, θα οδηγήσουν σε εκπλήρωση, σε επίτευξη των στόχων, θα χρειάζεται μια τακτική παρακολούθηση. Προβλέπει λοιπόν αυτό το πλαίσιο τα θεμέλια για την υλοποίηση ενός μηχανισμού παρακολούθησης. Ο μηχανισμός αυτός θα εξασφαλίζει ότι οι εθνικές στρατηγικές για τους Ρωμά υλοποιούνται, ότι οι πόροι οποίοι αποσκοπούν στην ένταξη των Ρωμά φτάνουν στον τελικό τους προορισμό και στους τελικούς δικαιούχους και ότι επιτελείται πρόοδος προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων για την ε, ένταξη των Ρωμά. Θα αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο σε αιτήσια βάση σε σχέση με την ένταξη των πληθυσμών ε, των Ρωμά στα κράτη-μέλη και πρέπει να σας πω ότι και το πλαίσιο το ευρωπαϊκό εδώ μας δίνει τη δυνατότητα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συσπηρωθούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και ο ευρωπαϊκός πληθυσμός ε, και η Ρωμά ειδικά πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για να μπει ένα τέλος στον αποκλεισμό 10 εκατομμυρίων συμπολιτών μας. Κάτι που δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε Ρέντινγκ. Τώρα δίνουμε το λόγο στον Επίτροπο Άντορ. Πρόεδρε, αξιότιμα οι βουλευτέ, η κοινωνική, η οικονομική κατάσταση των Ρωμά αποτελεί ένα θέμα προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την προηγούμενη μήνα εγκρίθηκε η έκθεση για ρούκα σχετικά με το θέμα αυτό και σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία ανακοίνωση για την εθνική στρατηγική ενσωμάτωση των Ρωμά και οι δύο αυτές εκθέσεις ε, συμβάλλουν στη συζήτηση για την αντιμετώπιση των Ρωμά και προετοιμάζουν και το επόμενο Συμβούλιο στις 19 Μαΐου που θα αφαιρεθεί αποκλειστικά στην ενσωμάτωση των Ρωμά. Τα έγκρα αυτά αποτυπώνουν την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναφερθούν και να αντιμετωπίσουν την κατάσταση ε, των Ρωμά που πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό. Τρία στοιχεία θέλω να θίξω. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις εθνικές στρατηγικές. Καταλαβαίνει ότι και αναγνωρίζει την πρωταρχική αιμοδιότητα των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Επίσης αποτυπώνει την βαθιά πεποίθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποτεχτεί ξενοφοβία, διακρίσεις, κοινωνικό αποκλεισμό, οποιοδήποτε είδους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηθικό αλλά και πολιτικό χρέος να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους με όλες τις πολιτικές και τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο σημείο. Ξέρετε ότι συμφωνήσαμε για μια συνεκτική στρατηγική για την ανάπτυξη ενός κοινωνικού μοντέλου με, με ε, ισορροπημένο τρόπο. Και χρειάζεται το απαραίτητο πολιτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση αυτού του α, ζητήματος. Θα πρέπει οι στόχοι 20-20-20 να ταχθούν και υπέρ του στόχου για την συμπερίληψη την ενσωμάτωση των ε, Ρωμά. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι βιώσιμο να αποκλίνονται τόσα εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να συνεχίσει ο αποκλεισμό των ε, Ρωμά στην Ευρώπη που ζούμε. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους στόχους για τη μείωση της φτώχειας ε, και για την εκπαίδευση αποτελούν βασικά ορόσημα για να προσμετρηθεί η ένταξη ενσωμάτωση των Ρώμα. Τέσσερις είναι οι τομείς οι οποίοι είναι στρατηγικής σημασίας για να ξεπεραστεί ο αποκλεισμός των Ρωμά. Πρόσβαση στην απασχόληση. Μεγάλο χάσμα μεταξύ να εξακολουθεί να, πρέπει, να υφίσταται μεταξύ των Ρωμά και των μη Ρωμά και θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους 20-20-20. Δεν θα τους πετύχουμε όμως αν δεν πετύχουμε τη συμπερίληψη των Ρωμά. Πρόσβαση στην εκπαίδευση. Θα πρέπει να μην υπάρχουν ε, ε, διακριτική μεταχείριση. Θα πρέπει όλα τα παιδιά να ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τουλάχιστον. Επίσης πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Και εδώ θα πρέπει να γεφυρωθούν τα χάσματα με, και να παρέχονται οι ίδιοι όροι στους Ρωμά. Και τέλος, πρόσβαση στην στέγαση και στις ε, βασικές ε, υπηρεσίες κοινή ωφέλειας. Η κατάσταση εδώ είναι πολύ χειρότερη για τους Ρωμά και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε κοινά αγαθά όπως ο ηλεκτρισμός και το νερό. Κατά τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δαπανίσει εκεί που πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει μια πρόταση για το πολιετές ε, πλαίσιο που θα ακολουθηθεί από συγκεκριμένε προτάσεις για τα διορθωτικά ταμεία. Θεωρώ ότι τα διορθωτικά ταμεία θα πρέπει να συνάδουν με την στρατηγική ε, για την Ευρώπη του 2020 και αυτό ισχύει για τους τομείς της πολιτικής για τους οποίους είμαι αρμόδιος για την απασχόληση και την κοινωνική συμπερίληψη αλλά και για την ε, ενσωμάτωση των Ρωμά θα πρέπει τα χρηματοπιστωτικά μέσα να καταστούν πιο αποδοτικά. Αυτό αποτελεί βασικό μου στόχο. Θα σταματήσω στο σημείο αυτό για να ακούσω και τα δικά σας σχόλια και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε, κύριε Άντορ. Το λόγο για το Συμβούλιο, ο ε, η Υπουργός, η κυρία Γκιόρη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, θα ήθελα να συνεχίσω στα αγγλικά. Η Ουγγρική Προεδρία καλωσορίζει την ανακοίνωση για το ευρωπαϊκό πλαίσιο, για την εθνική στρατηγική ε, ενσωμάτωση των Ρωμά. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το έργο σας, αλλά και για την προσωπική σας δέσμευση, Επίτροπε Ρέντινγκ, Άντρο και όλων εκείνων που συνεργάστηκαν για το πραγματικά σημαντικό αυτό επίτευγμα. Το στρατηγικό αυτό έγγραφο αποτελεί ένα τεράστιο βήμα για την πραγματοποίηση ενός από τους πιο σημαντικούς στόχους της Ουγγρικής Προεδρίας. Είμαι πεπισμένη ότι αν εγκρίνουμε αυτή τη σημαντική συμβολή για την βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των ΡΟΜ στην Ευρώπη σε συνδυασμό με το σχετικό ψήφισμα που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει της έκθεσης της Λίβιας για Ρόκα η ακραία ένδια και ο αποκλεισμό εξακολουθούν να απειλούν μεγάλες, ε, μεγάλο ποσοστό των Ρωμά στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να λέμε ότι είναι κρατικό το πρόβλημα αυτό και δεν μα αφορά. Επιπλέον, ο κόσμο ποτέ δεν μπορεί να θεωρείται, οι άνθρωποι ποτέ δεν μπορούν να θεωρούνται πρόβλημα. Όχι, αποτελούν μόνο μια ευκαιρία. Δεδομένη τη δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη, η προώθηση τη ενσωμάτωση των Ρώμα ανοίγει νέο δυναμικό το οποίο θα συμβάλλει στην αναπτυξή μας μακροπρόθεσμα. Η Ουγγρική Προεδρία πάντα πίστευε ότι πέρα από την καταπολέμηση των διακρίσεων που είναι απαραίτητη, χρειάζεται και ένα νέο μείγμα πολιτικών με τρία βασικά στοιχεία. Απασχόληση, εκπαίδευση και στέγαση. Οι ενσωματωμένες πολιτικές στους τομείς αυτούς και η σωστή εποπτεία της εφαρμογής τους από τα κράτη-μέλη και, από κράτη, και από την Επιτροπή θα κάνουν τη διαφορά. Οι προσπάθειες των κρατών μελών επίσης θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του 2020. Και όλα αυτά τα μέτρα μπορούν να ενσωματωθούν σε διάφορους ε, τομείς της πολιτικής. Τώρα αναγνωρίζουμε ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν επιπρόσθετη ευρωπαϊκή αξία. Και τι μέλη γενέστε τώρα. Η Ουγγρική Προεδρία σκοπεύει να παρουσιάσει και να συζητήσει την ε, ανακοίνωση στις 7 Απριλίου στην Σύνοδο στην Βουδαπέστη, στην οποία καλό ένθαρμα όσους το επιθυμούν να παρευρεθούν. Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης θα συζητήσει στις 12 Απριλίου το θέμα αυτό και μετά στις 19 Μαΐου το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ θα υιοθετήσει και τα ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου. Και επίσης στις 20 Μαΐου θα παρουσιαστεί στην Ουγγρική Προεδρία η σχετική έκθεση και στην, ε, στο Συμβούλιο ε, Γενικών Υποθέσεων στις 23 Μαΐου και τελικά τα αποτελέσματα αυτά θα εγκριθούν από το Συμβούλιο του Ιουνίου. Αυτό ασφαλώς δεν αποτελεί τίποτα παραπάνω παρά μια καινούργια έναρξη. Χρειάζεται συνεργασία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για να βοηθήσουμε αυτή την πραγματικά ευρωπαϊκή μειονότητα. Σας ευχαριστώ και τώρα ξεκινάμε τη συζήτηση με τους αγορητές των διαφόρων ομάδων. Ξεκινούμε με τον κύριο Τόκες για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμοι επίτρεπε. Ε, κυρία Γιαρόκα, σας ευχαριστούμε όλους που κάνατε ένα μεγάλο βήμα για την πραγματοποίηση της στρατηγικής ε, των Ρώμα. Στις 8 Απριλίου, την Παρασκευή, θα ξεκινήσει, θα, θα γιορτάσουμε την ε, Παγκόσμια ημέρα των Ρωμά. Θα συγκληθεί και για πέμπτη φορά η πλατφόρμα η Ευρωπαϊκή για τους Ρωμά Πρόκειται για πραγματικά ορόσημα. Πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο οποίο συμμετέχουν ωστόσο και λαμβάνονται υπόψη και οι τοπικοί φορείς. Ε, το ΕΛΚ εδώ και χρόνια ε, ζητά ένα τέτοιο σχέδιο δράσης για τη συμπερίληψη των Ρωμά και στις 24 Ιουνίου στην Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων ελπίζουμε να προκύψει μια πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρωμά, η οποία να μπορεί να λάβει και συνέχεια από πλευρά ανθρωπινών δικαιωμάτων. Πρόκειται για ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα, τα πιο ακραία προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Αποτελεί και ευθύνη όλων των κρατών μελών να διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών τους, να διασφαλίζουν το δικαίωμα ύπαρξης των πολιτών τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο όμως αυτό θα πρέπει να το τηρούν τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή η Στρατηγική για τους Ρωμά αποτελεί μια ένα τεχνικό ελάχιστο πρότυπο. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ωστόσο ότι αυτό το θέμα θα ενώσει όλες τις ομάδες και θα, θα καταστεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός. Και θα ήθελα να τονίσω κάποια σημαντικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής. Είναι σημαντικό ότι η ομάδα στόχος καθορίζεται βάσει όχι εθνοτικών κριτηρίων, αλλά οικονομικών κριτηρίων. Σημαντικό επίσης είναι ότι απαιτούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σημαντικό είναι η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των ευκαιριών, η εδαφική, ο εδαφικός αποκλεισμός. Είναι σημαντικό για να πετύχει το πρόγραμμα αυτό ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι κοινότητα των Ρωμά, οι εθνικές αρχές, προαπαιτείται μια στενή συνεργασία όλων αυτών των φορέων. Το θέμα αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολιτικές αντιπαραθέσεις, για την υποδάβληση α, μίσους, για στιγματισμό ομάδων. Όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά. Δεν είναι δυνατόν να ψάχνουμε συλλογικούς αποτυπωμένους τράγους το θέμα των Ρωμά στα πλαίσια της... μπορεί να επιληθεί στα πλαίσια των Ουγγρικών ταμείων που προτείνονται. Πρόκειται για ένα θέμα προτεραιότητας και ελπίζω να εγκριθεί το έγγραφο αυτό από την Σύνοδο του Ιουνίου. Σας ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές, η κυρία Φλασικόβα Μπενόβα έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ κυρία Προέδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα κύριε Επίτροπε να σας συγχαρώ καταρχάς που υποβάλατε το νέο πλαίσιο. Χαίρομαι που μετά από μακρές ε, διαπραγματεύσει ζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της ΠΙΕ υπογράφει αυτή την στρατηγική. Είναι καλή στιγμή διότι η κατάσταση γίνεται όλο και πιο σοβαρή. Πολλέ γυναίκε τώρα, μα και Ρώμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν αναξιοπρεπώς και είναι και θύματα τρομοκρατίας. Ε, στην Ουγγαρία έγινε κάποια τέτοια πορεία που τρομοκρατίες κατά τον Ρώμα στην Ουγγαρία και αυτό το δείχνει. Θα ήθελα να πω όμως και κάποια πράγματα που βρίσκω ότι δεν είναι σωστά. Δεν δέχομαι την απόψη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην διαβουλευτεί με τα δεμπλεκόμενα μέρη προετοιμάζοντα ε, το πλαίσιο. Είναι παράξενο λοιπόν από τη μία πλευρά το πλαίσιο να τονίζει ότι είναι σημαντική συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την ένταξη των Ρωμά, όμως ε, ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήθεσε σε διαβουλεύσεις με τους Ρωμά ή τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Όσον αφορά το περιεχόμενο, νομίζω ότι το πλαίσιο είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει αρμοδιότητε όσον αφορά το πανευρωπαϊκό αυτό πρόβλημα, όμω οι βασικέ αρμοδιότητε παραμένουν στα χέρια των κρατών μελών. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συντονίσει τι εθνικέ στρατηγικέ και να εξασφαλίσει τον έλεγχο, την εποπτεία των στρατηγικών. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να αναφέρουμε εδώ την εποπτεία των εθνικών στρατηγικών είτε έχουν τους ίδιους στόχους όπως οι ευρωπαϊκές στρατηγικές για να έχουν τους ίδιους στόχους όπως οι ευρωπαϊκές στρατηγικές. Σχετικά με αυτό πρέπει να πω ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έπρεπε να ακολουθήσει πιο σκληρή προσέγγιση όσον αφορά τις προσδοκίες που θα πρέπει να τίθενται από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν τέσσερι βασικοί τομεί που πρέπει να τονιστούν. Η εκπαίδευση, η απασχόληση, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση των Ρωμά. Ε, μαζί με συναδέλφου τη πολιτική μου ομάδα επισκεφθήκαμε κοινότητε τον Ρωμά στην Ευρώπη και είδαμε τα μάτια μα ότι αυτή είναι η βασική τομή που θα πρέπει να βελτιωθούν. Όμω θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτοί οι στόχοι αναφέρονται επίσης και στο πρόγραμμα της δεκαετίας για την ένταξη των Ρωμά. Τώρα ήρθε η στιγμή να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά. Ε, θα ήθελα να προσθέσω σε αυτούς τους τομεί άλλον έναν την καταπολέμηση όχι μόνο της διάκρισης αλλά της, των φραστικού ε, ρατσισμού και των πράξεων ρατσιστικής, ε, με ρατσιστικά αίτια. Η Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκάλυψε ότι έχουν, υπάρχουν ελλείψεις στα κράτη-μέλη όσον αφορά την χρήση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι γίνεται σωστή χρήση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να μειωθεί η γραφειοκρατία επίσης για τη χορήγηση των πόρων και θα πρέπει να επιτυχάνονται οι στόχοι προκαθορισμένοι. Ευχαριστώ εκ νέου, Επίτροπε, και συγχαρητήρια για την καλή δουλειά που κάνατε και ίσως να εκφράσω και μία ευχή το πρόγραμμα αυτό και το νέο πλαίσιο να δώσει θετικά αποτελέσματα που όλοι θέλουμε και επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Κυρία Φλασικόβα Μπενόβα, υπάρχει ένα γαλάζιο καρτελάκι σας ερώτημα του κυρίου Μπερμάιερ. Δέχεστε? Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, συνάδελφε Φλασίκοβα, που μου δίδατε την ευκαιρία να σας θέσω την ερώτηση. Ασχοληθήκατε με την έκθεση αυτή και ξέρετε τι προβλέπει. Ότι θα πρέπει να επιβάλλονται πρόστιμα από τα κράτη-μέλη αν υπάρχουν αποκλήσεις από την έκθεση ή αν υπάρχει απόκληση από τη στρατηγική. Τι πιστεύετε στην περίπτωση αυτή να πρέπει ένα κράτος να, να πληρώνει πρόστιμα αν δεν τηρείται υποχρέωση παρακολούθησης του δημοτικού, γιατί αυτό αποτελεί υποχρέωση σε κάθε χώρα. Αν ε, δεν συμβαίνει όμως αυτό, αν δεν, συμβαίνει, αν δεν παρακολουθούν τα παιδιά των Ρωμά το δημοτικό, θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν πρόστιμο στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι είναι καθήκον των γονιών να φροντίζουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. E, Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Μπενόβα. Να πω ένα πράγμα για αυτό που θέσατε. Είμαι υπέρ, υπέρ της ύπαρξης δικαιωμάτων, αλλά και συμμόρφωση πρέπει να υπάρχει με τις υποχρεώσεις. Είναι θέμα των γονέων, ρόλος των γονέων να προσέξουν τα πλευρά τα, συγγνώμη, τα παιδιά και τα δικαιώματά τους. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιτρέψουν τις δραστηριότητες και δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν ε, για τα λάθη των γονιών αν τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Ευχαριστώ. Για την Άλτε, Ήλτσεφ για δύο λεπτά. Ο κύριος Ήλτσεφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Γιαρόκα και τους εκπροσώπους ε, του Συμβουλίου της Ουγγρικής Προεδρίας για τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όταν μιλάμε για ένταξη των Ρωμά, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι αναφερόμαστε σε ένα από τα πιο επώδυνα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη χρηματοδότηση ε, και με νόμους κατά των διακρίσεων ή με προγράμματα ευαισθητοποίηση ε, τη κοινή γνώμη δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό μπορούμε να το λύσουμε μόνο με συνδυασμό και αυτών και πολλών άλλων προσεγγίσεων και όλα αυτά βέβαια με την απαραίτητη πολιτική βούληση. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα των εκατομμυρίων Ρωμά, που πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι Ούγγροι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι κτλ. Είναι άνθρωποι, είναι Ευρωπαίοι πολίτε. Έχουν τι ίδιε σίγουρα υποχρεώσει, αλλά έχουν και τα ίδια δικαιώματα και έχουν όμω περιορισμένε δυνατότητε. Πρέπει να ξεπεράσουμε κάποιε απερχιωμένε τάσει. Έχουμε λοιπόν πιθανότητες επιτυχία εάν ληφθούν ολοκληρωμένε δράσει πρωτοβουλίε από τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι δράσης ή ο αυτοσχεδιασμό θα είναι αντιπαραγωγικά, αλλά αναπαραγωγικές διαδικασίες. Ε, βέβαια, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές παρανοήσεις πολλές φορές γύρω από τους Ρωμά. Θα πρέπει λοιπόν με επαγγελματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, γιατί αντί ε, να αποσυναρμολογήσουμε και να αποσυνδέσουμε αυτή την μετακινούμενη, ε, την κινούμενη βόμβα, απλά θα τη μεταφέρουμε από το ένα σημείο στο άλλο. Όπως μεταφέρονται και αυτές οι κοινότητες. Ε, η στρατηγική είναι Σίγουρα μια προσπάθεια εκπαίδευση πολύ σημαντική. Πρέπει τα παιδιά των Ρωμά να μπαίνουν ε, και να φοιτούν στο σχολείο. Θέλουμε ε, επίσης ε, να περιορίσουμε τον αλφαβητισμό μεταξύ και των ενηλίκων Ρωμά. Και η Ρώμα βέβαια θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν και την κατάσταση διαβίωσης, όχι όμως μόνο πετώντας τους χρήματα. Σας ευχαριστώ για τους πρασίνους. Έχει το λόγο για δυόμιση λεπτά κυρία Φλότρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι καλά ναι αυτά σήμερα το ότι έχουμε για τους Ρωμά ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό που θα καταστήσει υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να γνωστοποιήσουν τη στρατηγική τους για την ένταξη των Ρωμά από τώρα μέχρι το τέλος του έτους Αυτές οι στρατηγικές θα αξιολογηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διεξαχθεί εκ νέου συζήτηση περίπου σε ένα χρόνο. Ξεκινά σήμερα λοιπόν ένας οδικός χάρτης που θα μας επιτρέψει, θα επιτρέψει εμάς τους βουλευτές στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στην κοινωνία των πολιτών να επαγρυπνούμε μονίμως όσον αφορά τους σημαντικότερους τομείς που παραθέσατε. Παρατηρώ ότι η έκθεση μάλλον ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνει υπόψη διάφορα σχόλια που διατυπώσαμε στην έκθεση του Κοινοβουλίου. Θα, αναφερθώ στην υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα εμπλέκεται στην αξιολόγηση στρατηγικών. Πιστεύω ότι αυτή η υπηρεσία δεν χρειάζεται να αποδείξει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που έχει στον τομέα και χρειάζεται και ανάπτυξη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης όσον αφορά την κατάρτιση δημοσιολαβητών που προέρχονται από την κοινότητα των Ρωμά. Είναι πολύ αποφασιστικό αυτό για να πετύχει το πρόγραμμα σε όλα τα επίπεδα. Και επίση, δίδεται προσοχή στους Ρωμά που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και η διάσταση της ε, διεύρυνσης λαμβάνεται υπόψη στην έκθεση και πιστεύω ότι ο καθορισμός κοινών δικτών για την ενίσχυση των μηχανισμών αξιολόγησης είναι κάτι απόλυτα ευπρόσδεκτο. Παρ' όλα αυτά στην ανακοίνωση θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις Πιστεύω ότι δεν αναφέρεται επαρκώς η ανάγκη της συμμετοχής των Ρωμά σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή της επεξεργασίας των προγραμμάτων, την εφαρμογή αυτών και την αξιολόγηση αυτών. Μιλάμε για ενημέρωση, μιλάμε για διαβούλευση εδώ. Χρειάζεται και η συμμετοχή της κοινότητας των Ρώμα. Είναι αποφασιστική σημασίας έχουν εμπειρία, καλές εμπειρίες, ε, καλά πειράματα που έχουν πετύχει στην Ευρώπη και αποδεικνύουν ότι εδώ υπάρχει μια δυναμία της ε, ανακοίνωσης. Δεύτερη δυναμία της ανακοίνωσης ότι αναφέρεται στη μη διάκριση οριζόντια σε κάθε από ένα από τους τομείς. Είναι πολύ σημαντικό θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει μια παράγραφος ειδική που θα αναφέρεται στην καταπολέμηση των διακρίσεων κατά της βίας, να αναφέρεται στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη της κοινότητας των, Ρωμά. Αυτή η πτυχή κατά των διακρίσεων θεμελιώδη δικαιώματα πρόσβαση στη δικαιοσύνη δεν αναφέρεται συγκεκριμένα ξεχωριστά και αποτελεί μια δυναμία του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μιλήσαμε για διαμεσολαβητές, πρόγραμμα που ξεκίνησε το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι καλό να αναφέρεται στην ε, ανακοίνωση. Θα θέλαμε επίσης να αναφέρετε και τις κατευθύντριες γραμμές που ήδη διατυπώθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ώστε να μην ακολουθούνται δύο στατηγικές ή δύο ήδη ε, βάσει αναφορά για την αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών. Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι θα ήταν ένα συν ε, στην ανακοίνωση. Τέλο, πιστεύω ότι η δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τελείωσε, ότι η ομάδα κρούση θα πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά τη, ούτω ώστε τα κράτη-μέλη καθημερινά να αισθάνονται την πίεση επάνω του Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την κοινωνία των πολιτών, και από πλευρά τη τοπική τοπικής για να εφαρμοστούν αυτοί οι προσανατολισμοί. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ο κύριος Κίρκοπ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Επιτροπή, η πρόταση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να ενσωματωθούν καλύτερα οι Ρωμά στα κράτη-μέλη και να βρεθούν τρόποι για να δοθούν ίσες ευκαιρίες και τα σωστά δικαιώματα στους Ρωμά. Το βασικό όνομα και βασικό στόχος ε, το, του εγγράφου θα πρέπει να είναι οι ε, ίσες ευκαιρίες και τα ίσα δικαιώματα. Ωστόσο, θεωρώ ότι όπως τα προηγούμενα προγράμματα είναι πάρα πολύ ε, βαριά η ατζέντα, πολύ φορτωμένη σε ό,τι αφορά οι αρμοδιότητες, τις αρμοδιότητες ε, των κρατών μελών σε θέματα στέγασης και εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνουν σεβαστές και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να καθορίζουν σχετικές πολιτικές. Ελπίζω ότι αυτή η στρατηγική θα αποτελέσει την έναρξη μιας νέας στρατηγικής, όπου καταρχάς θα ακούσουμε τους Ρωμά, γιατί ε, τα προγράμματα συνήθως είναι υπερβολικά περίπλοκα και δεν βοηθούν τους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Ε, δέκα χρόνια έχουν περάσει και σχεδόν τίποτα δεν έχουμε ε, πετύχει επί τόπου. Ελπίζω λοιπόν να είναι πιο εύκολη πλέον η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια και η εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύει χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να τα ξοδέψει με καλύτερο τρόπο πλέον. Ευχαριστώ για την ενωτική αριστερά. Για την ενωτική αριστερά, Ernst, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Αφενός είναι καλό να υπάρχει στρατηγική πλαίσιο για τους Ρωμά, αλλά αφετέρου θα πρέπει να βάλω νερό στο κρασί μου, γιατί αυτό που μας ε, ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, ε, φέρνει στις συζητήσεις μας με τους εκπρόσωπους των Ρωμά, οι οποίοι πάντα μας ε, ζητούσαν ακρίβεια στην στοχοθέτηση, σαφείς προδιαγραφές, συγκεκριμένες προδιαγραφές, σαφείς κυρώσεις σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, δεν, υπάρχει, δεν πληρούνται οι όροι αυτοί, αυτές οι προδιαγραφές. Ε, δεν υπάρχουν λοιπόν, υπάρχουν κενά, σαν ελβετικό τυρί είχαμε συμφωνήσει να είναι σαφής η στρατηγική, αλλά τι μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρα από σημεία αστίασης. Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία σε ό,τι αφορά για, παράληψη, για παράδειγμα τη λήψη αποφάσεων. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την επίτευξη των στόχων και αυτό που με εκνευρίζει ιδιαίτερα, είναι σκανδαλώδες, είναι ότι ρητά δεν αναφέρεστε τίποτα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της εχθρικότητας κατά τον Ρωμά. Λέτε ότι δεν χρησιμοποιείται τα διευθυντικά ταμεία για τους Ρώμα. Σας ρωτώ όμως ανοιχτά, δεν είναι μια αιτία για αυτό το γεγονός ε, η εχθρικότητα κατά τον Ρωμά. Εγώ το πιστεύω αυτό. Ε, εμείς από την ομάδα μου επικρίνουμε αυτή τη στάση. Θεωρούμε ότι δεν επαρκεί αυτό το έγγραφο και αναμένω τις σχετικές τροποποιήσεις του. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα... Για την Ευρώπη τη Δημοκρατία των Ελευθεριών έχει το λόγο για ένα λεπτό ο κύριο Μποργέτσιο. Ε, παρόλο που είμαι ευρωσκεπτικιστή, μπορούσα να θα υποστηρίξω μία τοποθέτηση για το 2020 για να αποφευθούν οι διακρίσει, οι δυσκολίε και η περιθωριοποίηση. Όμω χρειάζεται μια δράση αποφασιστική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον έλεγχο των συμπεριφορών των κρατών. Όταν αυτέ οι ομιλίε για το μεγάλο μέλλον, για το μεγάλο έλεγχο γίνονται από Ευρωπαίο Επίτροπο, εξακολουθεί να μην εξηγεί πώ στη χώρα του όμω στο μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου, αυτοί οι ομάδες που γύρω στη, μπορούν να εγκαταστούν στο σπίτι μου, στην Ιταλία, στη Γαλλία, με τα διάφορα εξαρτήματά του ενώ στο Λουξεμβούργο απαγορεύονται οι καταβλισμοί. Ε, λοιπόν, στην, ε, στη χώρα της κυρίας Ρέντινγκ δεν μπορούν καν να κατασκηνώσουν. Στη βασική ημερήσια εφημερίδα της χώρας μου, στην Κορία Ντελασέρα, ε, στη σημερινό φίλο λέει ένας πατέρας, ένας γονέας, δεν λέει το φίλο, πούλησε και συλλελήφθη στην Ιταλία διότι υπόλοιψε την κόρη του και πώλησε την κόρη του για να δοθεί στην ε, πορνεία. Άλλοι στέλνουν τα παιδιά τους να πάνε αλλού. Είναι εκείνοι που δεν τα παιδιά τους στο σχολείο παρά τις πιέσεις και την προσοχή των αρχών και των μεσολαβητών και των διαφόρων ενώσεων και φορέων. Θέλουμε να μιλήσουμε και για αυτά τα προβλήματα. Θέλουμε ε, να, ε, να μην θελοτυφλούμε και να δούμε ότι πολλά προβλήματα των ομάδων αυτών εξαρτώνται βασικά από αυτούς τους ίδιους. Τα προβλήματα των Ρωμά σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε με αυτό το σημείο. Οπότε πάμε στο επόμενο θέμα της μεσηδιάταξης. Έκθεση Φερνάντες